δημοκρατισμό. Άρα, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλω να απευθύνω χαιρετισμό προς αυτούς τους απεργού που υψώνουν το αίσθημα κατά αυτής της αδικίας. Κυρίες και κύριοι, έτσι ολοκληρώθηκαν και οι ομιλίες ενός λεπτού. Όλοι οι συνάδελφοι οι οποίοι είχαν ζητήσει το λόγο μπόρεσαν να παρέμβουν και ευχαριστώ τον ε, Επίτροπο. Σας εύχομαι καλή επιστροφή, καλό βράδυ. Αύριο το πρωί θα συνεχιστεί στις 8.30 το πρωί η συνεδρίαση και σας ευχαριστώ για την παρουσία σας.